Dear colleagues, welcome. Λοιπόν, σας καλωσορίζω. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή χρονιά. Ελπίζω να περάσατε καλά. Είμαστε εδώ τώρα για να συνεχίσουμε κοινή συνεδρίαση Econ και Budget Έχω επίσης τον κύριο Σαρφάμα αντιπρόεδρο της Budget για θέματα που έχουν σχέση με το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων. Δεν έχουμε πολλά να πούμε σε εισαγωγικά, εισαγωγικό επίπεδο. Εμείς πρέπει να κάνουμε μία αξιολόγηση για το ΕΦΣΙ. Αυτά όλα τα, κάνει, τα κάνουν οι δύο συνεισηγητές μας είναι σημαντικό και κρίσιμο θα έλεγα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας να υπάρξει μια επιτυχής βελτίωση των επενδυτικών μας σχεδίων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η προτινόμενη παράταση θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την περαιτέρω βελτίωση ε, των όρων που θα οδηγήσουν σε καλύτερες και περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάρβαμα αν θέλει να κάνει κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, ίσως κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη σαν παράδειγμα για τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Εγώ θα ήθελα να πω εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ότι δεν συνεδριάσαμε από το Νοέμβριο του 2015 για τα θέματα αυτά, αλλά ταυτόχρονα όμως κάναμε τρεις αξιολογήσεις, πήραμε τρεις αξιολογήσεις από την Επιτροπή για το σύστημα εγγυήσεων, τη λειτουργία του ΕΦΣΥ και την εκ των υστέρων αξιολόγηση και είχαμε επίσης και την εξωτερική αξιολόγηση των Ernst Young για τη λειτουργία του Ταμείου. Υπήρξαν και άλλες προτάσεις. Ε, πήρε απόφαση στις 6 Δεκεμβρίου επ' αυτόν το Συμβούλιο. Τα πράγματα είναι γνωστό έχουν και θα συζητήσουμε σήμερα το πώς θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Ας περάσουμε στην ουσία λοιπόν. Οι δύο εισηγητές, η Μπούλμαν ή η Φερνάντες, ένας από τους δύο. Κύριε Φερνάντες, σας ευχαριστώ, θέλω να σας συγχαρώ όλους. Να ευχηθώ φυσικά σε όλους καλή χρονιά. Να ευχηθώ Χρόνια πολλά και στα ευρωπαϊκά όργανα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Νομίζω ότι τα 550 εκατομμύρια κατοίκων της Ένωσης έχουν ανάγκη αυτές τις ευχές και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε ε, επιτυχία σημαντική το Ταμείο αυτό. Αυτό θα το πετύχουμε βελτιώνοντας όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του FC. μέχρι τώρα με τις εμπειρίες που έχουμε μπορούμε να κάνουμε μια θα έλεγα περιγραφή των προβλημάτων τα οποία έχουν υπάρχουν. Υπάρχει ένα περιθώριο περαιτέρω επενδύσεων πάνω από 240 δις ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, βρισκόμαστε ε, πέραν των προσδοκιών μας 388.000 χιλιάδες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από το ΕΦΣΥ και ο αριθμός του συνεχίζει να αυξάνεται. Το Ταμείο αυτό εφαρμόζεται πλέον και λειτουργεί και στις 28 χώρες αντίθετα με το παρελθόν όπου υπήρχε ένας πιο περιορισμένος αριθμός. Πάνω τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο γρήγορα στους άλλους τομείς όσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ και ένα, ενάμιση χρόνο το θέμα που είχε τεθεί είναι αν το Ταμείο αυτό και ο τρόπος που λειτουργεί έχει επιπτώσεις αρνητικές θετικές εννοώ ε, στην πραγματική οικονομία. Και η πρόταση που γίνεται τώρα είναι να περάσουμε από το 315 δις που ήταν η αρχική πρόβλεψη στα 500 δις. Ήδη ε, ένα μεγάλο ποσό έχει κινητοποιηθεί. Θα πρέπει όμως ε, να έχουμε περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας για να δούμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του επενδυτικού αυτού ταμείου στον τομέα της απασχόλησης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε ανάγκη μεγάλη για περαιτέρω επένδυση έτσι ώστε να καλύψουμε τα ρήγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Και γι' αυτό ακριβώς λοιπόν το Ταμείο αυτό είναι σημαντικό. Τέθηκε και το θέμα της προσθετικότητας. Ε, εδώ υπάρχουν δυσκολίες για την βελτίωση της κατάστασης. Αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των προγραμμάτων θα πρέπει να ερμηνεύσουν με σωστό τρόπο την έννοια του όρου. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει και αυτή να κάνει μια καλή θα έλεγα ερμηνεία του όρου και οι υπηρεσίες της να κατανοήσουν το τι καλύπτει ο όρος προσθετικότητα στο σύνολό του. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει συστηματικά θα έλεγα το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσουμε και μια γεωγραφική ισορροπία. Έχουμε βέβαια να κάνουμε με ένα ταμείο το οποίο δεν έχει σαν βασικό στόχο την αντικατάσταση του Ταμείου Συνοχής. Το ταμείο αυτό θέλει να λειτουργεί εκεί όπου η αγορά είναι ελληματική και να στηρίξει προγράμματα που δεν στηρίζονται με άλλους τρόπους. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρξει υπερσυγκέντρωση γεωγραφική, δεν πρέπει να υπάρξει υπερσυγκέντρωση θεματολογική και θα πρέπει να λειτουργήσει το Ταμείο αυτό έτσι ώστε οι χώρες μέλη και οι περιφέρειές τους να ωφεληθούν. Θα πρέπει επίσης το Ταμείο αυτό να λειτουργεί με προληπτικό τρόπο και να χρησιμοποιηθεί για στόχους στρατηγικής. Εδώ είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε δώσει την απαιτούμενη προσοχή. Πρόκειται για την πλατφόρμα συμβουλών προς τους επενδυτές, το EIPP. Ε, εδώ απαιτείται να λειτουργήσουν καλύτερα αυτές οι διαδικασίες και θα πρέπει επίσης να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας και σε σχέση με τα ελάχιστα ποσά τα οποία μπορεί να χορηγούνται ε, υπάρχουν συνδυασμοί βέβαια ανάμεσα σε διάφορες χώρες και ανάμεσα σε διάφορους τομείς. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν και πλατφόρμες διμερείς επενδυτικές ανάμεσα στις ε, διάφορες χώρες. Σαν παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας οι πλατφόρμες αυτές μπορούν να ομαδοποιήσουν τις επιμέρους ε, προτάσεις έτσι ώστε να καλύψουν το κατώτερο ποσό πέρα από το οποίο η ε, παρέμβαση του Ταμείου είναι εφικτή. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν βελτιώσεις που οφείλουμε να κάνουμε βγάζοντας καταρχάς τα, τα σωστά συμπεράσματα για την εκτέλεση και λειτουργία του Ταμείου αυτού μέχρι τώρα. Είναι συνολικά θετική η λειτουργία του. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Ούντο Μπούλμαν, εισηγητή από την Επιτροπή. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρη. Ευχαριστώ και εσάς Χωσέ Μανουέλ για τα εισαγωγικά λόγια. Και από τη δική μου πλευρά εύχομαι σε όλες και όλους καλή καινούργια χρονιά με καινούργια ενέργεια και καινούργιο θάρρος. Άλλωστε, καλό ξεκίνημα για το νέο έτος είναι και αυτή εδώ η συζήτηση για νέες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί και επεποίθηση μεγάλης πλειοψηφίας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η νομοθεσία που έχει θεσπιστεί ως τώρα είναι ορθή. Ωστόσο, όπως είπε και ο Χωσέ Μανουέλ, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με όλα όσα αφορούν την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και σε ό,τι αφορά την επιλογή των έργων και το ζήτημα της προσθετικότητας που αναφέρθηκε πριν. Διότι υπάρχουν και έργα τα οποία θα είχαν χρηματοδοτηθεί ούτως ή άλλως και χωρίς το εύση. Καλύψαμε πράγματι κάποια κενά με στρατηγικές επιλογές. Η απάντηση συχνά είναι όχι. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία για να αναπτύξουμε τις ε, επενδύσεις. Η απάντηση πάλι είναι όχι. Υπήρξαν αρκετές επενδυτικές πλατφόρμες για να μεταφερθούν οι πρωτοβουλίες στις περιφέρειες και να ενισχυθούν ιδίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως για μικρά ή και ακόμα πιο μικρά έργα και να δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν εξυγχρονιστικές δραστηριότητες. Και εκεί λίγα πράγματα έχουν γίνει. Κάτι άλλο είναι το ζήτημα της οργανωτικής δομής του ΕΦΣΙ. Και αυτή πρέπει να μας απασχολήσει. Συχνά μας προκαλείται η εντύπωση ότι ο βασικός φορέας που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το παρακάνει με το business as usual. Το παρακάνει μέσα στις γνωστές παραδοσιακές δομές και με τα γνωστά κριτήρια επιτυχίας και δεν εγκύπτει αρκετά σε αυτό το αναγκαίο πνεύμα καινοτομία, το οποίο πρέπει να διέπει τι πρωτοβουλίε και του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των χωρών μελών. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της ΕΦΣΙ 2.0 που μας έχει διαβιβάσει περιλαμβάνει θετικά πράγματα. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τα δεδομένα του βαθμολογίου, του scoreboard. Επίσης, η προσπάθεια να επιτευχθεί ένα υψηλότερο κβάντουμ επενδύσεων για περιβαλλοντικά έργα. Το άλλο είναι το ερώτημα πώς μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερο αποτέλεσμα χωρίς περισσότερα χρήματα. Είναι και αυτό ένα χρήσιμο ερώτημα. Να γίνουν προσπάθειες δηλαδή να αυξηθούν οι επενδύσεις, αλλά πρέπει να αυξηθεί, ε, αυξηθεί η αποδοτικότητα των επενδύσεων. Το Ευρωκοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία τάσεται υπέρ της παράτασης της ισχύω του ΕΦΣΥ. Δεν μπορούμε όμως να υπογράφουμε απλώς χωρίς να επιφέρουμε διορθώσεις στα όσα μας φαίνονται προβληματικά. Θα επενδύσουμε σε αυτή την νομοθεσία όπως κάναμε άλλωστε και με το FC 1.0, έχουμε μπροστά μας ε, δύο πράγματα ανοιχτά. Την έκθεση αξιολογήσεως, που θα πρέπει πρώτα να εγκύψουμε σε αυτήν, γιατί θέλουμε να δούμε ποια πράγματα πήγαν καλά, ποια λιγότερο καλά ή ποια χρειάζονται διόρθωση. Και μετά έχουμε και την ομοθεσία για το fc 2. Θα τα προχωρήσουμε αυτά και θα τα εντάξουμε το ένα μετά το άλλο στην ε, προσπάθειά μας και θεωρώ ότι μέχρι μέσα Μαΐου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πορεία τους μέσα από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ώστε να καταλήξει μετά η νομοθετική διαδικασία, όπως ελπίζω, εντός του εξαμήνου της Μαλτέζικης Προεδρίας και πριν από τις θερινές διακοπές. Αυτό είναι με απλές αδρές γραμμές το χρονοδιάγραμμά μας. Θα καθορίσουμε όσο γίνεται νωρίτερα το χρονοδιάγραμμα για τις συναντήσεις και εμπειρογνώμονες διότι το ΕΦΣΙ έχει και πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, γνωρίζετε ποιες είναι και οι, ε, είναι μάλλον και οι διοικητικοί περιορισμοί, οι γραφειοκρατικοί αν θέλετε περιορισμοί εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο, δηλαδή ότι οι επιτροπές δεν μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν άπειρο αριθμό συνεδριάσεων ανά εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και τα πράγματα που μας είχαν απασχολήσει ήδη με το FC1 και θα πω στον Χωσέ Μανουέλ ότι έχουμε λάβει πολλή υποστήριξη και διακομματικά με πολλή δέσμευση από πολλούς, με πολύ επικοδομητικό πνεύμα από μέλη πολλών και ποικίλων κομματικών ή μάλλον πολιτικών ομάδων, νομίζουμε ότι ο στόχος τα αξίζει όλα αυτά. Και σας ευχαριστώ ήδη από τώρα για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος του Κάρας. Εύα, εσείς έχετε το λόγο λοιπόν εξ ονόματος του κύριου Κάρας. Χαίρετε προς όλες τις κατευθύνσεις. Είμαι Ότμαρ Κάρας απόψε ο οποίος κολλείται σήμερα διότι έχει σημαντική συνάντηση στην Βιέννη. Μιλώ λοιπόν ε, για λογαριασμό του. Λέγει λοιπόν ο Τμαρκάρας ότι αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να κοιτάξουμε προς τα πίσω στα όσα ήδη έχει επιτύχει το EFCI. Πιο σημαντικό ωστόσο να κοιτάξουμε προς τα εμπρός, στο μέλλον και να δούμε ποια πράγματα μας αναμένουν τα επόμενα χρόνια. Επειδή ο κανονισμός EFCI βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού σχεδίου επενδύσεων του Προέδρου Γιούνκερ και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει αρχίσει να ισχύει εδώ και μία διετία και από τότε έχει επιτύχει σημαντική αύξηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και θετικά ως αφετηρία. Επιθυμώ να προσθέσω κάτι σχετικά με τους αριθμούς που ανέφεραν και άλλοι προηγουμένως. Ως τώρα έχουν κινητοποιηθεί 164 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή δισεκατομμύρια ευρώ, ε, δηλαδή το 52% του ε, προβλεπόμενου ποσού και έχουν ενισχύσει πάνω από 200 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν προσελκύσει και φρέσκες επενδύσεις που είναι αναγκαίες παντού. Βρισκόμαστε λοιπόν στη σωστή τροχιά. Όμως μένει πολλή δουλειά ακόμη να γίνει και οι τρεις αξιολογήσεις, κάποιες από αυτές αναφέρθηκαν ήδη, οι Ernst και Young έχουν καταδείξει πολλές ε, ελλείψεις στην εφαρμογή του EFCI που πρέπει βέβαια να τις εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Οι νομοθετικές προτάσεις του Σεπτεμβρίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν τις, ε, τα κενά αυτά. Ταυτόχρονα υπάρχουν και μένουν ανοιχτά αρκετά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προκλήσεις όπως η ανάγκη της ξεκάθαρης προσθετικότητας των έργων για να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες της αγοράς ή κάποιες καταστάσεις που δεν είναι άριστες, high risk profiles, η κλίμακα του ποσοστού της συμμετοχής στις πλατφόρμες επενδύσεων που ακόμα δεν έχουν εμφαρμοστεί και η συνεργασία με εθνικές τράπεζες αναπτύξεως. Ο συνάδελφος μου πακάρας επιθυμεί να καταστεί απόλυτα σαφές και για όσους παρακολουθούν από το διαδίκτυο ότι οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αγώνας 100 μέτρων, είναι μαραθώνιος και γι' αυτό χρειάζεται μακρά πνοή και σε έργα υποδομής και σε καινοτομίες όπως νέες ενεργειακές πηγές και το ψηφιακό μας μέλλον. Είμαι βέβαια, ή βέβαιος μάλλον, ότι θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά επιτυχώς καθώς και άλλα θέματα τα οποία κρεμούν στους επόμενους μήνες και πάλι ε, για λογαριασμό του Ότμαρ ευχαριστώ και τους δύο συνεισηγητές για την θαυμάσια ως τώρα συνεργασία. Και αν με επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ακόμη ένα λεπτό να πω τη δική μου προσωπική άποψη, διότι είμαι σκιώδης συζηγήτρια της ΙΜΚΟ για τη γνωμοδότηση. Πολύ σύντομα λοιπόν, εγώ λέγω πάντοτε ότι η FCI δεν αποτελεί πανάκια για όλα μας τα προβλήματα ε, των επενδύσεων στην Ευρώπη, όμως αποτελεί ένα εργαλείο που διευκολύνει και που έχει αποδώσει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ένα πολύ σημαντικό ε, θέμα το οποίο θέσαμε στη γνωμοδότησή μας της Επιτροπής ΥΜΚΟ και που θα ήθελα πολύ οι υπεύθυνοι συγκητές που είναι σήμερα παρόντες εδώ να συμπεριλάβουν στην έκθεσή τους ε, την ιδέα αυτή. Βρήκαμε ότι μόνο 10% των επενδύσεων του FSI στον ψηφιακό τομέα είναι μόνο 10%. Άρα είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτός. Και όλοι οι συνάδελφοί μου στην ΕΜΚΟ, σας παρακαλώ, ε, θα πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει ο πρόεδρος Γουαρθιέρη. Μάλιστα, μάλιστα. Ενώ χρειάζονται για να προωθηθούν οι επενδύσεις ε, σε αυτές ε, τις επενδύσεις που έχουν υψηλό κίνδυνο αλλά και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Από, με το δικό μου όνομα λοιπόν θα εργαστώ και εγώ πάνω στην πρόταση EFI 2.0. Ευχαριστώ πολύ. Από τους Σοσιαστέ και δημοκράτες έχουμε κάποιον. Για στο όνομα του Έντερ. Α, ο κ. Μάρκα, εσείς μάλιστα. Κύριε Μάρκα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το EFSI έχει σχεδιαστεί για να χρηματοδοτεί επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Αυτά ακριβώς είπαν και οι συγητές μας. Πρόκειται για συμπληρωματικέ επενδύσεις δηλαδή, οι οποίες ποτέ δεν θα γίνονταν χωρίς την βοήθεια του EFSI. Συνεπώς, το επενδυτικό αυτό ταμείο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό σε βάρος του ορίζοντα 2020, του, της συνδέοντα συνδέοντας την Ευρώπη κλπ. Τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν για αυτά τα προγράμματα. Και το λέω ότι αν τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιούμε και τα χρησιμοποιούσαμε για παράδειγμα στη Γαλλία για τα σπίτια που επλήγησαν από τις πλημμύρες ενώ σε άλλες χώρες αντίστοιχες ανάγκες χρηματοδοτούνται από τον εθνικό προπολογισμό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστό. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ του να έχουμε προγράμματα τα οποία βελτιώνουν την ενεργειακή μας αποτελεσματικότητα, αλλά θα πρέπει να είναι και συμπληρωματικά. Η προσθετικότητα δηλαδή θα πρέπει να οριστεί σαφώς, γιατί μερικές φορές κάνουμε πολύ καλά προγράμματα όπως αυτό στη Γαλλία, αλλά τα χρήματα φερούνται από άλλα προγράμματα. Και καλό είναι επί της ουσίας να έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα αυτά εκεί, αλλά θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί αυτά και από τον Εθνικό Προπολογισμό. Τώρα, για το δεύτερο στάδιο του επενδυτικού αυτού ταμείου, που επικεντρώνεται στις περιφέρειες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους τομείς που έχουν αγνοηθεί μέχρι τώρα. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην παίρνουμε χρήματα από προγράμματα καινοτομίας και από άλλους τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σάντερ Λούνς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους σας για το 2017. Τώρα, για το ΕΦΣΥ. Για το πρώτο στάδιο του παιδιτικού αυτού ταμείου είπαμε ότι η μόχλευση των χρημάτων για να αυξηθούν οι επενδύσεις είναι μια θετική προσέγγιση. Όμως τονίσαμε επίσης ότι δεν πρόκειται και για το μαγικό ραβδί όσον αφορά τις επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνονται μεν στην Ευρώπη, αλλά σιγά σιγά και επικρατεί ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα στην αγορά και θεωρούν πάντα ότι είναι ένας ακριβώς τρόπος για να κάνουν business. Εμείς πάντα υπογραμμίζουμε τα βασικά, ότι δηλαδή αν θέλουμε μακροπρόθεσμα να έχουμε επενδύσεις πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Λιγότερη γραφειοκρατία, να μειωθούν τα εμπορικά εμπόδια και να φροντίσουμε οι χώρες μέλη ότι εφαρμόζουν τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και για μένα αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά, εξακολουθεί να είναι ένα χώρο που δεν έχει ασφάλεια όσον αφορά τις επενδύσεις. Πάντως για την ανταλλαγή αυτή απόψεων θέλω και κάποιες ερωτήσεις να θέσω. Λοιπόν, υπάρχουν, μάλλον να δώσω κάποιες απαντήσεις. Ναι, υπάρχουν θετικά σημάδια στην αρχική περίοδο όσον αφορά το EFSI, αλλά δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ήδη από τώρα την πραγματική επιτυχία. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι για να έχουμε περισσότερες επενδύσεις δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε τόσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Οπότε ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και τώρα έρχομαι στις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την αξιολόγηση και μετά για την προσθετικότητα. Για την αξιολόγηση. Η ανάλυση έχει γίνει πραγματικά θα περιοριστούμε σε αυτές τις τρεις ε, αξιολογήσεις ή θα ζητήσουμε κι άλλες. Και όσον αφορά το συνδέοντας την Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020, τι έχει γίνει, έχει βελτιωθεί καθόλου εκεί η κατάσταση και με την καινοτομία. Δεύτερον τώρα, προσθετικότητα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Εδώ πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει τους στόχους της Οικομισιόν, αλλά από άλλα χαρτοφυλάκια μπορούμε να κρίνουμε πραγματικά το ΕΦΣΥ. Να δούμε κατά πόσο τα προγράμματα είναι πραγματικά βιώσιμα, αυτά που χρηματοδοτούνται δηλαδή, και κατά πόσο θα είχαν υλοποιηθεί εκτός του ΕΦΣΥ όχι. Η προσθετικότητα θα πρέπει να οριστεί πιο συγκεκριμένα στις διάφορες χώρες μέλη. Και τελειώνω με μία ακόμα ερώτηση επί του περιεχομένου. Θα βοηθούσε να δούμε το θέμα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις ε, επενδυτικές τράπεζες. Κατά πόσο τηρείται ή όχι δέος επιμέλεια. Είναι θέματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Bernd Κόλμερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα βεβαίως ε, καλή χρονιά σε όλες και όλους και μακάρι να τα καταφέρουμε καλύτερα από ό,τι τον προηγούμενο χρόνο. Ασφαλώς είναι καλό να καθίσουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις επενδύσεις, άρα την οικονομία και εν τέλει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Για τέτοια ερωτήματα όμως πρώτα-πρώτα πρέπει να ξεκινούμε, κατά τη γνώμη μου, από το ερώτημα είναι ιστορικά ή επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το κράτος με άμεσες επενδύσεις ή με τέτοιες έμεσες χρηματοδοτήσεις μακροπρόθεσμα έχει ποτέ ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα ή εν τέλει την ζημιώνει, κάτι που πιστεύω εγώ ότι γίνεται. Ούτε είμαι και τόσο θαραλέος όσο οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου που είπαν έως τώρα ότι είναι πολύ πεπισμένοι από τις επιτυχίες του EFCI. Αυτές τις επιτυχίες ως τώρα δεν είδα πουθενά να αξιολογούνται. Θα πρέπει ε, πράγματι να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Εάν επιθυμούμε να προωθήσουμε επενδύσεις στον δημόσιο τομέα των χωρών μελών της Ένωσης, αυτό σημαίνει ότι ενθαρρύνουμε τις χώρες αυτές να δανείζονται για να επενδύουν. Μα αυτά δεν χρειάζονται το εύση, μπορεί να γίνουν μια χαρά και χωρίς το εύση. Στον ιδιωτικό δε τομέα πιστεύω ότι καμιά αρχή δεν μπορεί να υπάρξει όσο καλά οργανωμένη και να είναι, που να τα καταφέρει να ρυθμίσει όλες εκείνες τις αναγκαίες λεπτομέρειες που θα εξασφαλίσουν την προσθετικότητα των έργων και αυτά μακροπρόθεσμα να μπορούν να στηριχθούν στα πόδια τους, μόνα τους. Αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε με πάρα πολύ κριτικό πνεύμα πριν να λάβουμε οποιασδήποτε αποφάσεις. Κύριε Σάρβαμα, εσείς τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και που τηρήσατε τον χρόνο σας. Θα παρακαλέσω όλους τους και όλους να ε, τηρήσουν το όριο των ε, δύο λεπτών. Και μην θυμιλισμονείτε ότι έχουμε κάτι άλλο μετά στις 6 ώρα. Μην ξεπεράσουμε λοιπόν τον χρόνο μας. Ε, η φιλελεύθερη, η ομάδα Άλντε, ε, επιθυμεί κάποιον να λάβει τον λόγο. Έχετε κάποιον σκιώδη συγητή παρόντα. Αν όχι, τότε θα προχωρήσουμε στον κύριο Τούρβολτς για δύο λεπτά, που είναι ο σκιώδης των ε, προπολογισμών της Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους. Κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου διαλύματος ε, μελέτησα την ευρωπαϊκή ιστορία. And one of the most interesting points with... Α, διάβασα τη βιογραφία του Ζαν και τα απομνημονεύματα. Μετά τον πόλεμο ήταν ε, επίμονος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε να επενδύσουν το 27% του ΑΕΠ τους για να μπορέσει να ξεκινήσει η Ένωση. Έχουμε μείνει λίγο πίσω λοιπόν σε σχέση με το απαιτούμενο ποσοστό και αυτό οδηγεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και ο Μπούλμαν και ο Φερνάντες ε, έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε στην παρούσα φάση είναι <clears throat> η λεγόμενη τεχνική προσθετικότητα, δηλαδή εάν θέλουμε να δίνουμε σε μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις χρήματα, και σωστό είναι αυτό, τότε στην ουσία θα οδηγηθούμε σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι επιχειρήσεις αυτές τελικά θα μείνουν πίσω, δεν θα κάνουν τις απαιτούμενες κινήσεις μόνες τους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε σχέση με την ε, προσθετικότητα σε θέματα τεχνολογίας. Αν το καταφέρουμε αυτό, τότε νομίζω θα έχουμε πετύχει ένα σημαντικό βήμα και η Ευρώπη θα έχει καλύψει την ε, απαιτούμενη προσπάθεια. Πολύ σημαντικό, αναφερθήκατε και στο Ζαμονέ και μείνατε πάνω, κάτω από το 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα. Ο Ντεμάζη έχει το λόγο. Καλή χρονιά και από μένα. Η συζήτηση αυτή δεν διεξάγεται μέσα σε κενό αέρος, αλλά μέσα σε μια βαθιά κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό θα προχωρήσω λίγο περισσότερο σε βάθος. Δεν είμαι και τόσο ευνηδιασμένος που ορισμένες πτυχές του ΕΦΣΥ δεν ε, προχωρούν τόσο καλά όσο παρουσιάζουν ορισμένοι. Αυτή η story ότι το βασικό πρόβλημα είναι η απέχθεια στον κίνδυνο στην Ευρώπη δεν με πείθει, διότι στο παρελθόν είχαμε και υψηλότερες επενδύσεις και πριν από την κρίση. Και είναι σχετικά προφανές ότι μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο όπου περικόπηκαν οι δημόσιες δαπάνες η όθηση για επενδύσεις είναι περιορισμένη. Νομίζω λοιπόν ότι μια πρόθεση για το νέο έτος, μια καλή πρόθεση για το νέο έτος θα πρέπει να είναι και πώς θα προωθήσουμε τις δημόσιες επενδύσεις. Και με, δεν με εκπλήσει όταν διαθέτει κανείς μια τέτοια εγγύηση στους ιδιώτες επενδυτές ότι προσελκύονται και ότι η προσθετικότητα δεν είναι βεβαίως ε, εγγυημένη διότι ό,τι μου προσφέρουν δωρεάν το παίρνω και φεύγω. Τώρα λοιπόν που θα επανεξετάσουμε ολόκληρο το οικοδόμημα θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά. Έχουμε και τις κοινοπραξίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως τη γερμανική Bundesbank, όπου εκεί και το ανώτατο ε, ε, ε, ομοσπονδιακό δικαστήριο κατέληξε ότι τελικά είναι υψηλότερο το κόστος για τον φορολογούμενο, διότι συγχρηματοδοτούμε με τον τρόπο αυτό και το κέρδος των, ιδιωτών επενδυτών. Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε μήπως πρέπει να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό στις επενδύσεις. Δημόσιες επενδύσεις αυτές, οι δημόσιες επενδύσεις δε, να εξαιρεθούν από τα κριτήρια του ελλείμματος. Τα πράγματα αυτά τα συζητούμε και για τους εξοπλισμούς, για την άμυνα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για τις δημόσιες επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Α, είστε εδώ. Ωραία. Εσείς έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, εδώ είμαι και εγώ εύχομαι καλή χρονιά σε όλου. Θα είμαι σύντομη. Θέλω όμω να επικεντρωθώ στις ε, κοινωνικές και ε, συνεταιριστικές τράπεζες. Προσπαθώ να έχω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επ' αυτού, αλλά δεν τα καταφέρνω έχει γίνει ένα πολύ περίπλοκο σύστημα και για τους απλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε χρήματα από εκεί. Εμείς μιλάμε για απλοποίηση, λέμε να υπάρχει διαφάνεια για τους πολίτες μας. Ναι, θέλουμε να προωθήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να τις βοηθήσουμε να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια αυτά, στην Ιρλανδία για παράδειγμα, αλλά δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες, η μία πάνω στην άλλη που προστίθεται. Οπότε, πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το σύστημα, δεν το βλέπω εγώ. Και μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια μέχρι το 2016 εγώ δεν έχω δει συγκεκριμένα στοιχεία από αυτού. Οπότε για άλλη μια φορά είναι οι ιδιωτικοί επενδυτέ οι οποίοι υποφελούνται. Και δεν είμαστε κατά των επενδύσεων, όχι. Αλλά έχουμε αποτύχει όσον αφορά την κοινωνική οικονομία και εξακολουθούμε σε αυτήν την αποτυχία. Τα χρήματα αυτά δεν είναι προσβάσιμα σε αυτούς που περισσότερο τα χρειάζονται. Οπότε να προσέξουμε πάρα πολύ καλά την αξιολόγηση αυτή. Χρειαζόμαστε αυτέ τι πληροφορίε, χρειαζόμαστε τι επιπτώσει, χρειαζόμαστε διαφάνεια και λογοδοσία. Και μα ε, εγγύθηκαν ότι θα τα έχουμε στην αρχή. Δυστυχώ όμω δεν τα έχουμε. Δεν έχουν ε, όλες οι χώρες τα συστήματα αυτά δημοσίων ε, τραπεζών, δηλαδή για παράδειγμα. Και σας λέω, ο κόσμος μερικές φορές δεν ξέρει καν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχουν μοντέλα α, β, γ. Συζητάμε για απλοποίηση, ναι, αλλά ας αφήσουμε στην πάντα τη ρητορική και ας περάσουμε στην πράξη ρεαλιστικά για να βοηθήσουμε αυτούς που περισσότερο έχουν ανάγκη. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος και ο εισηγητής από την ε, ΕΚΟΝ, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ και εγώ στέλνω τις ευχές μου για καλή χρονιά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι αυτή τη χρονιά θα δουλέψει και πάνω στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μέχρι τώρα η αξιολόγηση του ΕΦΣΥ καταλήγει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επιτυχές, πρέπει να συνεχίσει. Τελεία και παύλα. Μα αυτή δεν είναι μια αξιόπιστη αξιολόγηση. Αν κοιτάξουμε τις διάφορες ανεξάρτητες αξιολογήσεις που έχουν γίνει υπάρχει Υπάρχουν πολλές επικρίσεις. Εμείς στηρίξαμε το πρώτο στάδιο του επενδυτικού αυτού ταμείου, γιατί θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι είναι ζωτική σημασία οι επενδύσεις. Ναι, αλλά πώς πρέπει να δούμε ε, πού βάζουμε τις προτεραιότητες, πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει διαφάνεια. Όλα αυτά τα θέματα έχουν δεχτεί επικρίσεις και από εσωτερικέ αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και από τον κύριο Ντεγιόν και από άλλους που έχουν κάνει αξιολογησεις της ευρωπαικη τραπεζα επενδυσεων αλλα και απο τον κυριο ντεγιον και απο αλλου που εχουν κανει αξιολογησει τετοιες και από το γραφείο του Ντεγιάν κτλ. Οπότε, ναι, θέλουμε να συνεχίσουμε με επενδύσεις, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε με καλό τρόπο, έτσι ώστε οι επενδύσεις αυτές να πηγαίνουν εκεί που πρέπει και ότι η ταξινόμηση που γίνεται, η ιεράρχηση των επενδύσεων γίνεται με το σωστό τρόπο και μα στο υποσχέθηκαν αυτό με το σχέδιο Juncker. Αυτό θέλουμε να έχουμε. Πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Το να συνεχίσουμε ε, και να μην αλλάξουμε τίποτα δεν θα λειτουργήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλά θα κάνει να πει και κάτι παραπάνω, αντί να λέει είναι πρόγραμμα Juncker, οπότε όπως και να έχουν τα πράγματα είναι επιτυχές. Μα αν θέλουμε να κοιτάξουμε σωστά, πρέπει να κοιτάξουμε την κατεύθυνση που παίρνουν οι επενδύσεις. Και ακόμα πολλές επενδύσεις για τις μεταφορές, για παράδειγμα, πηγαίνουν στα ορυκτά. Μα είναι προς τη στραβή κατεύθυνση αυτές, ε, ε, αυτό. Αν δείτε επίσης τη γεωγραφική κατανομή, το Ηνωμένο Βασίλειο παίρνει πάρα πολλές ε, επενδύσεις και η Γαλλία, η Γερμανία. Μα δεν είναι εκεί που λείπουν οι επενδύσεις κυρίω Και τρίτον, απασχόληση. Και εδώ θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μα το κριτήριο αυτό. Στις μέχρι τώρα αξιολογήσεις είδαμε ότι μόνο με στέλνει θέση απασχόλησης είναι λίγο πολύ 7.000. Που είναι πάρα πολύ μικρό το νούμερο αυτό. Πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν η ιεράρχηση, η διαφάνεια και να υπάρχει διαφάνεια και στο βαθμολόγιο για να μπορεί το κοινό να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Αν αυτά δεν αλλάξουν, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε εμείς, εντάξει, θα συνεχίσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα, ώστε οι επενδύσεις ε, αυτές να γίνονται βάσει μιας καλής επενδυτικής πολιτικής που θα αλλάξει τα πράγματα. Ευχαριστούμε κύριε Έκχαουτ λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μαραγάλ δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Θέλει εκείνος εκ μέρου των Πρασίνων. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση φυσικά να αντικαταστήσω τον κύριο Μαραγκάλ, ποιος είναι στην Ισπανία. Με το FDD έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο δεν τον ακούμε καλά τον ομιλητή. Έχω φωνή που ακούγεται και δεν χρειάζομαι το μικρόφωνο. Λοιπόν, το θέμα είναι πόσο θα επιβαρυνθούν οι πολίτες φορολογικά και οι επιχειρήσεις ε, οι οποίες αναγκάζονται να υποκύπτουν σε αυτά τα οποία αποφασίζουν οι υπάλληλοι και οι γραφειοκράτες που δεν ξέρουν από επενδύσεις. Νομίζω ότι πράγματι οι πολιτικές αυτές ε, σε καμία περίπτωση δεν έχουν την επιτυχία την οποία μας είχαν υποσχεθεί ότι θα είχαν και ακόμα και αν υπάρχει κυβερνητική έγκριση θα έλεγα των προγραμμάτων αυτών, τότε αυτό δεν αρκεί έτσι ώστε να γνωρίζουμε την ποιότητα των προγραμμάτων αυτών και φυσικά τα προγράμματα αυτά θα αποτύχουν όπως ακριβώς και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Νομίζω ότι πρόκειται εδώ για κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ευτυχώς που εμείς θα φύγουμε από την Ένωση, οπότε δεν θα έχουμε τέτοιου προβλήματα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, λέει ο κ. Σταβάρμα. Δεν βλέπω κάποιον άλλο από τον προϋπολογισμό, γι' αυτό δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο του ΙΕΝΕΦ για την ΕΚΟΝ. Όχι, δεν θέλει το λόγο. Καλώς. Παίρνει το λόγο ο κ. Γκουαλτιέρη. Περνάμε στο Κατστιάι λοιπόν. Ο κύριος Ρούμπικ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Και εγώ θα υποστηρίξω και πάλι ότι χωρίς παραγωγή, χωρίς υπηρεσίες δεν μπορεί να υπάρξει κατανάλωση. Όποιος θέλει λοιπόν να είναι κοινωνικά δίκαιος πρέπει να φροντίσει να υπάρχει παραγωγή και παροχή υπηρεσιών. Και για την παραγωγή χρειάζονται επενδύσεις και όποιος δεν είναι βέβαιος ότι όσα επενδύουν, επενδύει καταλήγουν σε επιτυχία, οφείλει να πράξει έτσι ώστε να γίνουν επιτυχία. Και αυτό σημαίνει και κάποια διάθεση ανάληψης κινδύνου. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να δούμε τι κάνουμε με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ιδίω όσες ανταγωνίζονται στην παγκόσμια αγορά. Βεβαίως και χρειάζονται εγγυήσεις. Έχουν να δώσουν έχουν, χρειάζονται εγγυήσεις για να μπορούν ε, να προχωρούν και σε εξαγωγέ. Και γι' αυτό μιλούμε για χρηματοδότηση. Όπου τα χρήματα του δημοσίου των χωρών μελών είναι πολύ περιορισμένα. Γι' αυτό και πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν δισεκατομμύρια. Αυτά θα πρέπει να τα διαθέσει τα πρώτα δηλαδή χρήματα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις χώρες μέλη, κάτι το οποίο θα οδηγήσει και σε χαμηλά επιτόκια και επομένως σε σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης και στο Emission Trading System μπορούν και εκεί τα χρήματα που θα εισπραχθούν να προβλεφθεί ότι θα διατεθούν ιδίω για το EFCI, EFSI, συγγνώμη ώστε να επιτευχθεί και εκεί μεγαλύτερο αποτέλεσμα μόχλευσης. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Γιατί θα σημάνει ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Αν μπορέσουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι και τα έργα αυτά επενδύσεων για τις επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να αναλυθούν και αυτές, δηλαδή οι εγγυήσεις για τις επενδύσεις αυτές, από το Ταμείο EFSI. Αυτό θα είναι μεγάλο όφελος και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές για αυτό το σημαντικό θέμα. Πολλά ακούστηκαν μέχρι τώρα. Θα ήθελα όμως να βεβαιωθούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα έλεγα συμμετέχουμε στην διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Να πω ότι την τελευταία φορά είχαμε τρει ξεκαθαρου δυο δύο-τρεις ξεκάθαρους στόχους και ήταν πολύ σημαντικό να διευκρινηθεί η θέση του Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχει ήδη ξεκαθαρίσει λίγο το πεδίο. Ευτυχώς η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά κάποιο τρόπο λαμβάνει πολλές από τις δικές μας θέσεις υπόψη για το FC1, θέσεις οι οποίες δεν είχαν στην απτική φάση ληφθεί υπόψη όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τους δύο αρχικούς εισηγητές εδώ. Πάνω σε αυτό έχουν υπάρξει κάποια επιμέρους στοιχεία τα οποία έχουν υπογραμμιστεί και τα οποία είναι προφανή και δεν θα επιμείνω. Η οικολογική μετάβαση σαν παράδειγμα. Μήπως θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτήν την ιδέα η οποία είχε, είχε συζητηθεί αλλά στο τέλος δεν έδωσε θα έλεγα ένα ποσοστό, μια ποσόστοση επαρκή. Και επίσης το θέμα της στήριξης της πλατφόρμες. Ένα σημείο στο οποίο, δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να επιμείνω και είναι δύο σημεία άξονες θα έλεγα για τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Το πρώτο, στην αρχή είναι σαφές ότι δεν ήμασταν 100% όλοι πεπισμένοι ότι η διαχείριση του ταμείου αυτού θα έπρεπε να γίνει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είδαμε ότι βασικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε κάποιος άλλος να κάνει τη δύσκολη δουλειά. Από την άλλη ε, θα έλεγα τέθηκε ε, σε συζήτηση το θέμα της ικανότητας διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της άποψης που έχει για το τι συνιστά ε, σύγχρονη επένδυση σήμερα. Έχει να κάνει βήματα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως προς αυτό και αυτά τα βήματα θα πρέπει να γίνουν πριν ξεκινήσει το FC2. Είναι υποχρεωμένη να λάβει περισσότερους κινδύνους, αυτό πρέπει να τις το θυμίσουμε. Και σε σχέση τώρα με τις κοινωνικές επενδύσεις, είναι το δεύτερο σημείο. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι ο πυρήνας των ανησυχιών γενικά όταν μιλάμε για το Ταμείο Γιούνκερ. Αλλά νομίζω ότι όπως είπε και ο συνάδελφος από την ομάδα των Πρασίνων έχουν γίνει σημαντικές εργασίες ιδιαίτερα ε, με την όφηση του Λάσλο Άντορ, του τέος Επιτρόπου Κοινωνικών Υποθέσεων, που επιμένουν στην χρήση του Ταμείου Ιούνκερ για την προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων και αυτό βρίσκομαι ότι είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει να το στηρίξουν σαν κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κυρία Μπερές. Δεν έχω κάποιον άλλο που έχει ζητήσει το λόγο. Ε, δεν υπάρχει πλέον άλλος ο οποίος έχει ζητήσει το λόγο. Συνεπώς έχουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Καζόνη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την ευκαιρία που δώσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο σε αυτή την πρώτη σας συνάντηση. Όπως είπατε και όπως είπαν και πολλά άλλα μέλη, η εφαρμογή του ευσύ από πλευράς μας θεωρείται αρκετά επιτυχής. Οι στατιστικές έχουν ήδη δοθεί για να το στηρίξουν, δεν θα τις επαναλάβω τώρα. Ε, ε, δείχθησαν τα ποσοστά τα οποία καλύφθηκαν και ε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομική βάση που μπορούμε να φτάσουμε. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πάβει να είναι ενήμερη κάποιων σημείων κριτικής που ακούστηκαν όπως επίσης και κάποιων σημείων ανεπάρκειας οι οποίες ήρθαν στην επιφάνεια στα πλαίσια της λειτουργίας του ΕΦΣΥ. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στο θέμα της προσθετικότητας είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας, γιατί από τη μία στη νέα μας πρόταση εμείς προσπαθούμε να είμαστε πιο πιστοί σε αυτά τα οποία έχει πει το Κοινοβούλιο και μένουμε στο θέμα της προσθετικότητας λέγοντας ακριβώς που θα πρέπει να σταθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας σε σχέση με τα κοινά της αγοράς στον τομέα της χρηματοδότησης, με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα. Ταυτόχρονα και εδώ αντιχωρισμένες από τις παρατηρήσεις που έγιναν σήμερα εδώ, η η πρόταση για εξαίρεση επενδύσεων στους αυτοκινητοδρόμους και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να καλυφθεί καλύτερα από τις αγορές. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να πούμε ότι η προσθετικότητα δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα επιβληθεί με βάση άκαμπτα κριτήρια και κανόνες. Είναι ένα θέμα κυρίως διαφάνειας και δύο σημαντικές πλευρές στον συγκεκριμένο τομέα είναι πρώτον η ανάγκη που υπάρχει ε, και την οποία υπογραμμίζει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητά από την Επενδυτική Επιτροπή να μας δώσει εξηγήσει γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ωφεληθεί από τις εγγυήσει του κοινοτικού προϋπολογισμού και από την άλλη από τη δημοσιοποίηση του scoreboard, του πίνακα αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συνολικά θα βελτιώσει τους όρους προσθετικότητας. Επίσης συνειδητοποιούμε τις ανάγκες που υπάρχουν για την βελτίωση της περιφερειακής και γεωγραφικής ισορροπίας της εφαρμογής του ΕΦΣΥ. Εδώ θα πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο ε, το hub το λεγόμενο, το κέντρο ε, χορήγηση συμβουλών το επενδυτικό ε, και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κέντρο αυτό, η πλατφόρμα αυτή ε, τα περιφερειακά αντίστοιχα κέντρα και εθνικά κέντρα συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων. Οι επενδύσεις δεν γίνονται με αυτόματο τρόπο και γι' αυτό απαιτείται χρόνος για τη σωστή προετοιμασία και χρόνος για τη συλλογή σωστής ενημέρωσης. Ταυτόχρονα για τις χώρες συνοχής εμείς προτείνουμε κάποια ε, πλέον ευέλικτα κριτήρια επιλεξιμότητας. Επιτρέπουμε για τις χώρες αυτές σαν παράδειγμα την χρηματοδότηση των οδικών υποδομών, αυτοκινητών δρόμων μάλλον. Και επίσης ε, να μην ξεχνάμε ένα σημαντικό θέμα, το θέμα της εύκολης συνεργασίας με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και εδώ υπάρχει και η πρόταση Omnibus για τον κανονισμό. Υπάρχουν και κάποια άλλα ποιοτικά σημεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα οποία εν έχουν προέλθει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς πράγματι όπως είπε και η κυρία Μπερές λάβαμε υπόψη αυτά τα οποία μας είχατε πει. Είναι σημαντικό για μας να αποφύγουμε σαν παράδειγμα την πλευρά αποφυγής πληρωμής φόρου που πολλές φορές μπορεί να βγει μέσα από το Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές, να ευχαριστήσω φυσικά τον κύριο Φερνάνδες που μας έδωσε μια καλή εικόνα της κατάστασης και με τον κύριο Μπούλμαν με τον οποίο ίσως δεν συμφωνούμε απολύτως σε σχέση με την κατάληξη των διαπραγματεύσεων πριν το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε όμως γρήγορα έτσι ώστε να συνεχίσει και το FC αμέσως μετά το καλοκαιρινό ε, διάλειμμα. Σας ευχαριστώ κύριε Κασόνη. Τώρα περνάμε στον τελευταίο γύρο των συνεισηγητών για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Ο κύριος Μπούμακ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. θα συνοψίσω τις παρεμβάσεις των συναδέλφων, τους οποίους και τις οποίες ευχαριστώ. Θεωρώ ότι μπορούν να συνοψιστούν ως εξή οι παρεμβάσεις τους. Ορισμένοι συνάδελφοι λένε κατά βάση δεν βλέπουμε ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και ότι αν πάει να αναμειχθεί το κράτος όλα θα γίνουν χειρότερα. Υπεραπλουστεύω βέβαια. Γνωρίζω την συζήτηση αυτή την έχουμε διεξαγάγει και επί χρόνια πολλά και σε βάθος εδώ στην ε, παρούσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν λέω ότι είναι λάθος να γίνει η συζήτηση αυτή, λέω ότι δεν είναι σημαντικό να γίνει. Ε, μάλλον δεν λέω και ότι δεν είναι σημαντικό, λέω ότι είναι σημαντικό να γίνει. Αλλά εν ώψη της υψηλής ανεργίας σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν ώψη των σημαντικών γνωστών άλλωστε ελλημάτων και στην οικονομία και στην διοίκηση, στα ψηφιακά και ούτω καθεξής. Το θεμελιώδες ερώτημα για μένα έχει ήδη επιληθεί από την εποχή του Αδάμ Σμιθ 1767 και ο οποίος είχε αγωνιστεί για μια ανάμειξη του κράτους μέσα σε ένα παραγωγικό ρόλο και μάλιστα ήταν προδημοκρατική η προσπάθεια αυτή πριν από την σύγχρονη δηλαδή, δημοκρατία. Ήθελε να θεσπίσει ένα κρατικό μονοπόλιο και οδήγησε σε μια ιδέα εν τέλει οικονομικής διαμόρφωσης, διάρθρωσης που είναι αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Νομίζω ότι η άποψη πλειοψηφίας των επιτροπών μας είναι ότι μπορεί κανείς να συνδυάσει εφιώς την κρατική πρωτοβουλία με την ιδιωτική πρωτοβουλία και μπορεί να τα καταστρέψει και μπορεί να την κάνει τόσο ανόητα ώστε και μια χώρα μέλος που έχει τις υψηλότερες εξαγωγές να μην μπορεί να επισκευάσει τους αυτοκινητοδρόμους της να υπάρχουν χώρες οι οποίες να μην ξέρουν τι να κάνουν την ηλιακή ενέργεια, την ενέργεια του ανέμου και του νερού. Εάν μπορέσουν να τα φτιάξουν όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ευφυή προσπάθεια συνδυασμού μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Και νομίζω ότι αυτό απηχείται και στις περισσότερες παρεμβάσεις των συναδέλφων, που όμως από την άλλη πλευρά διαπιστώνουν ότι υπάρχουν και ελλείμματα. Για παράδειγμα, ελλείμματα στην κοινωνική πολιτική. Ελλείμματα εφαρμογής, διότι δεν επιλέγουμε επαρκώς ή δεν είναι αρκετά ποιοτική η επιλογή που κάνουμε. Ή το ζήτημα ότι η τεχνολογική συνιστόσα υποτιμάται μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών επιλογής. Το γεγονός ότι πρέπει να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, η governance, ότι όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν ταχύτατα στην έκθεση αξιολογήσεως και ότι γι' αυτά πρέπει να βασιστούμε στις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει από την εφαρμογή του EFSI 1 και να προσαρμόσουμε το νέο EFSI ώστε να φτάσουμε σε ένα πιο ποιοτικό καθεστώς ποιοτικών επενδύσεων. Ελπίζω να έχω την ε, συναδελφική σας υποστήριξη και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την συνεργασία. Σας ευχαριστώ κύριε Μπούλμαν. Ο εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέρφους. Υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο και θα συνεχίσει να είναι ενωμένο εφόσον οι δύο συνεισηγητές βρίσκονται στο ίδιο πνεύμα και οι σημερινές παρεμβάσεις αυτό ακριβώς ε, έδειξαν ότι έχουμε τον ίδιο στόχο. Με το ΕΦΣΥ καταφέραμε να μειώσουμε κατά ένα δις το κόστος από τον ορίζοντα 2020 και την ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Βελτιώσαμε και το κείμενο γιατί διαπιστώσαμε την ανάγκη καλύτερης ε, διαχείρισης. Επίσης αναφερθήκαμε και στην εδαφική συνοχή και στη δημιουργία απασχόλησης. Θα συνεχίσουμε όμως να έχουμε ένα πρόβλημα, ότι το ταμείο αυτό απαιτεί δράση από τους συμμετέχοντες, από τις περιφέρειες. Έδωσα ένα παράδειγμα, την Ενεργειακή Ένωση. Αυτή χρειαζόμαστε. Μιλάμε για αυτήν. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι χώρες μέλη έχουν την υποχρέωση να δράσουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εκείνο το οποίο είπε ότι οι γείτονε χώρε μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγγύηση για το στόχο αυτό. Ναι, αλλά οι χώρε μέλη πρέπει να μιλάνε μεταξύ του. Πρέπει οι χώρε μέλη να χρησιμοποιούν τι πλατφόρμες μεταξύ χωρών για το στόχο αυτό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως στο γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε σήμερα. Ο στόχος της σημερινής συνάντησης ήταν να δούμε κυρίως την εφαρμογή, τη χρήση. Αρχίζουμε όμως να μιλάμε και για το μέλλον και είναι καλό αυτό. Θεωρώ ότι το κοινωνικό σκέλος, η γεωργία, η αλία, οι δατοκαλλιέργειε είναι μέσα στον κανονισμό αυτό, είναι στο πνεύμα του κανονισμού. Μπορούμε να τα διατυπώσουμε με περισσότερη σαφήνεια, εντάξει. Μπορούμε να έχουμε πλατφόρμες για τον κοινωνικό τομέα με τον κανονισμό που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Πρέπει επίσης να επιμείνουμε και για έναν άλλο στόχο. Και αυτός είναι ότι οι πλατφόρμες αποτελούν το μέσο το καλύτερο για να συγκεντρώσουμε εθελοντική δράση. Για να βάλουμε τα προγράμματα μαζί, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από αυτό το ταμείο, αλλά και τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Χρειάζεται αυτή η συνύπαρξη. Επενδυτικό ταμείο και διαρθρωτικά ταμεία, με καλό συντονισμό. Έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα εφόσον χρησιμοποιήσουμε μαζί τα μέσα αυτά που διαθέτουμε. Έχω και μια άλλη ανησυχία και αυτή είναι ότι γνωρίζουμε τα προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί. Γνωρίζουμε τα προγράμματα τα οποία έχουν απορριφθεί με μια ρήτρα εμπιστευτικότητα. Δεν ξέρουμε όμω ποια είναι τα προγράμματα αυτά τα οποία δεν έχουν μπει καν στο σύστημα. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πολλέ φορέ λέει είναι πολύ μικρό το πρόγραμμα που προτείνει, δεν μπαίνει καν μέσα στο σύστημα. Και όμως θα ήταν σημαντικό να δούμε ποια είναι τα προγράμματα εκείνα που οι δικαιούχοι θα θέλανε να χρηματοδοτήσουν, αλλά δεν μπαίνουν καν στο σύστημα. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξέρω και τον ε, εξαίρετο συνεισηγητή που συνεργάζεται μαζί μου, τον Νούντο Βούλμαν, από τη δικιά μας την πλευρά λοιπόν θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να έχουμε τον κανονισμό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Με την ε, τωρινή τη Μαλτέζικη Προεδρία. Ελπίζω να υπάρξει ίδια φιλοδοξία και από τα άλλα θεσμικά όργανα. Από τη δικιά μας την πλευρά είμαι σίγουρος. Το έχουμε δείξει και κατά το παρελθόν ότι μπορούμε να δουλέψουμε γρήγορα και να συνεργαστούμε με όλους. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να συνεισφέρουν όλοι, όλες οι πολιτικές ομάδες, γιατί ο στόχος ε, καλύτερης ε, ανταγωνιστικότητας και επενδύσεων, απασχόληση, εδαφική συνοχή, όλα αυτά είναι στόχοι κοινοί μεταξύ μας. Η Ευρώπη, αν ρωτάτε, χρειάζεται επενδύσεις, βεβαίως και χρειάζεται επενδύσεις. Η Ευρώπη έχει αδυναμίες στις αγορές, ναι, θα πω σε αυτή την ερώτηση, market failure, πράγμα που σημαίνει ότι το χρειαζόμαστε αυτό το ταμείο και χρειαζόμαστε και περισσότερη απασχόληση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας. Είμαι σίγουρος ότι μαζί θα τα καταφέρουμε. Θα καταφέρουμε να έχουμε ένα βελτιωμένο κανονισμό και μετά πάντα θα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ότι θα πρέπει να τηρούμε τον κανονισμό, να ερμηνεύουμε σωστά τον κανονισμό, τον οποίο είμαι βέβαιος ότι θα εγκρίνουμε σύντομα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ακούσαμε τον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Φερνάντες, και όντως πολύ σωστά λέει ότι υπάρχει ε, συμφωνία μεταξύ μας και το ότι θέλουμε να εργαστούμε γρήγορα με τη συμμετοχή όλων. Η ταχύτητα δεν ε, έρχεται σε αντίθεση με την ποιότητα του έργου μας. Οι συνεισηγητές μας θέλουν ε, πρώτα την αξιολόγηση, μετά το νέο κείμενο. Έχουμε εδώ και το χρονοδιάγραμμα. Θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε και μήπως μπορούμε να κάνουμε το χρονοδιάγραμμα κάπως πιο σφιχτό, δεν ξέρω. Θα το συζητήσουμε. Ίσως να είναι ναι. συμβατό το χρονοδιάγραμμα αυτό, προκειμένου να καταλήξουμε επί Μαλτέζικης Προεδρίας. Και ο Χωσέ Μανουαλ Φερνάντες πολύ σωστά είπε ότι το νομοθετικό κείμενο είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, αλλά επίσης σημαντική είναι και η καλή χρήση των ε, μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, των εργαλείων αυτό. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ό,τι και αν αλλάξει, πάντα υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουμε την πρακτική, το μείγμα, ας πούμε, του ΕΦΣΥ με τα διαρθρωτικά ταμεία, την χρήση των διαφορών πλατφορμών, τη χρήση της προσθετικότητας και επενδύσεις που ίσως δεν έχουν γίνει λόγω αυτού που είπαμε market failure. Αυτό το νομοθετικό έργο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να βελτιώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ε, ρύθμιση στο τρέχον στάδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Λοιπόν, οι ημερομηνίε είναι οι 23 Ιανουαρίου κρόση, 25 Ιανουαρίου στη συνέχεια για την εφαρμοστική έκθεση. Μετά έχουμε 13 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο, προθεσμία για τις τροπολογίες 28 Φεβρουαρίου, υποβολή της νομοθετικής έκθεσης 15 Μαρτίου. Εδώ είναι που βλέπω, δεν ξέρω αν θα το τηρήσω θα δούμε. Τέλος πάντων, μπορούμε να κερδίσουμε μια εβδομάδα. Ανταλλαγή απόψεων 3 Απριλίου επί των ε, τροπολογιών, 10 Απριλίου στη συνέχεια και 15 Μαΐου ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και 17 Μαΐου αρχίζει ο τριμερής διάλογος. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να τελειώσουμε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και να έχουμε εγκρίνει την νομοθεσία τότε. Ο συμπρόεδρός μου εδώ μήπως έχει να προσθέσει κάτι. Ναι, ίσως πάρα πολύ σύντομα θέλω να προσθέσω ότι παρόλο που κατανοώ βέβαια απόλυτα το τι προσπαθούμε να κάνουμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που δεν είναι ένα άλμα αλλά ένας μαραθώνιος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, παρόλα αυτά θα έλεγα ότι όλοι πρέπει να επιδείξουμε κριτικό πνεύμα. Γιατί αυτό που το χείρμα στο οποίο μπαίνουμε είναι πραγματικά ένας μαραθώνιος. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο και στο μεταξύ όλοι γνωρίζουμε ότι το πολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη δεν δείχνει να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό πολύ φιλικά. Οπότε να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Πρόεδρος, καλώς. Έτσι ολοκληρώνουμε την συνάντησή μας. Η επόμενη συνάντηση κοινή εκόνο προπολογισμη 23 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα για το ίδιο αυτό θέμα, έτσι. Ωραία, έληξε η συνεδρίαση αυτή.